Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε την ψηφοφορία μας. Έχετε λάβει και τον κατάλογο, τους καταλόγους των ψηφοφοριών στα εγγραφά σας, ανά πολιτική ομάδα. Και ξεκινάμε λοιπόν με τη δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πάτε λοιπόν τις ε, κάρτες σας, βάλτε τις μέσα, στις, τις μέσα εδώ στα μηχανήματα. I ask you very simple question. Και σας ερωτώ, σας αρέσει να ψηφίζετε στις, ε, τις Δευτέρες 4 ώρα το μεσημέρι. Καταβούληση ο Πρόεδρος. πέρασε της πληροφορίας. Δεν είναι ε, πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Μάλλον κάποιοι από εσά βγάλατε τις κάρτες και δεν θέλατε να ψηφίσετε. 32 συνάδελφοι ψήφισαν, καταπληκτικός αριθμός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Άδειε του συναδέλφου Άντρα Γκιούρκ ό,τι αφορά την σταδική της Ευρωπαϊκή Ένωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση αερίου. Τροπολογία 56 ψήφι υπέρ. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω λοιπόν και πάλι. Συγητή Άνδρα Γκιούκ. Ε, θέμα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αγροποιημένο φυσικό αέριο και αποθήκευση αερίου. Α ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία, συνάδελφοι. Τροπολογία 56 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. NV1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Αφέτε 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφετ 2 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν για την ΑΦΕΤ 2. Πέρα τη υποφορίας απορριπτεται απορρίπτεται. NV3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είτε ένα τμήματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά ε, για να ελέγξουμε την 73 λοιπόν ψηφίζουμε για την 73 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 πνευματική ψηφοφορία πρώτο μήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή NV5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 τραν υπέρ, κατά, αποχές για να ελέγξουμε λοιπόν για την τραν 5. Απορρίπτεται. Να κλείσουμε όμως πρώτα την ψηφοφορία. Όχι, γίνεται δεκτή, δεν απορρίπτεται. Δεκτή. Ε, ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό να ελέγξουμε. Συμβαστική δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αποχές δεκτή. 96 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε λοιπόν την 96. Ελέγχουμε την 96. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 τραν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 121 υπέρ, 121 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 121. Πέραση της φοφορίας απορρίπτεται. Τραν 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρουμε. Ξανά. 32 τραν υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Α, όχι, είναι δύο μαζί. 126 και 127 λοιπόν. Ψηφίζουμε από κοινού. Γιατί είναι ίδιε. 126 και 127 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε λοιπόν την 131. Πέραση της φοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 μαζί με την 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές Δεκτεί 140, 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ κατά ας ελέγξουμε. Την 162. I close Πέρας. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Ξανά. Παρακαλώ να την αλλάξουμε. 163 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 164 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 α μαζί με την προηγούμενη ήταν 190 και 191 είναι ταυτόσιμες και απερίφθησαν η τροπολογία 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 επέ κατά αποχές. Ορίστε. Θέλετε έλεγχο, παρακαλώ. Ναι, 193. We vote 193. Ψηφίζουμε την 193 πέρα. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Ορίστε. Όχι, 197. Λάθος. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Μαζί με τη 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά έλεγχος χρειάζεται εδώ παρακαλώ ψηφίσουμε την τροπολογία 215 I close the vote. Rejected. Πέρας τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, δεν είδα καλά. 14 έμβη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2-16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.30 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 23 ε, είναι τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 6 της ΑΦΕΤ υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. ΑΦΕΤ 11 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η 14α υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για τη συμβαστική 14 α. 14α. Πέρας. Απερίφθη. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. Οι τέσσερα των μεταφορών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ σε 2.44 the Πέρας. Απορρίπτεται. Είναι τα δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να σηκώνετε χέρια, δεν σας βλέπω. Είναι τα δύο. Η τροπολογία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρασε. Μην κρίνετε. Σας προκαλώ να σηκώνετε χέρια. Είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε, Είναι τα 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.42 υπέρ, κατά. 2.42 παρακαλώ να το ελέγξουμε. Άνοιξη η ψηφοφορία, κλείνει. Απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 18 της NV υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για 18 της Επιτροπής Περιβάλλοντος NV. Πέρας. Απορρίπτεται είναι το 9 σε τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η άφετ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές ΕΝΒΙ NV12 υπέρ, κατά. Ας το ελέγξουμε και αυτό. 12 λοιπόν της ΕΝΒΙ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 16 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 της ΕΝΒΙ υπέρ. Κατά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 κατά ελέγξτε παρακαλώ 14 της Επιτροπής Μεταφορών. Transport Πέρας. 15 των μεταφορών υπέρ. Against. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζητώ συγγνώμη, θέλει έλεγχο αυτό. Δεν τα χέρια, τι να σας κάνω. 16 των μεταφορών. Έλεγχος. Πέρασε. Mm. Αγκρίθηκε. Ε, πού να τους μαντέψεις. 2,58 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2,59 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τραν το μεταφορών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές έλεγχος είναι η τροπολογία παριθμών 20 την οποία και ελέγχουμε πέρας Απορρίπτεται. Η συμβαστική 17α υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη συμβαστική 17α. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το πρόγειο 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίψονται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίψονται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. την 28 επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 31. Παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 36. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 39 υπέρ. Against. Abstention accepted. 40 in favor. Against. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ να ελέγξουμε τις 44 ηλεκτρονικά ελέγχουμε τις 44 check. We will see. I, I close the vote. Accepted. Accepted. I said rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε επιπρόσθετα προς την συμβαστική 18, η τροπολογία 45, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 51. I close the vote. Rejected. rejected. Uh, compromise Απορρίπτεται. Συμβεστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 3 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται 4 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 ε- πηδάμε στην 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Συγγνώμη, η 11. Υπέρ, από την 9 ναι, πάμε στην 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ 16. Συγγνώμη, ζητάει ο Πρόεδρος. Περνάμε στην 16 λοιπόν. Τροπολογία 16 πέρα. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά 16. I close the vote. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές να ξαναελέγξουμε να ψηφίσουμε για άλλη μια φορά 17 ήταν αυτή λοιπόν πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε γκρίθηκε συγχαρητήρια στον εισηγητή και ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη δεύτερη λίστα ψηφοφορίας ε, σχέδιο γνωμοδότησης ε, επί της πρότασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακή φορτότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά. Κάρλος Ζωρίνιο είναι ο εισηγητής. Συμβεβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 111 ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 111 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συγγνώμη, 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ 131 να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 131. Ελέγχουμε την 131 πέρας ψηφοφορίας. Το ίδιο με πριν έγινε. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 138. 139 συγγνώμη με 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ 145 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 145. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβεστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεστική 3 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 36. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά. Υπέρ, συγγνώμη, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ας ψηφίσουμε την 53 ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 53 δεν φαίνεται καθαρά πέρας ψηφοφορίας ε, εγκρίνεται καθαρά 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 5 τροπολογία 5 ελέγχουμε Πέρας ψηφοφορίας. Σαφώς έγκρινεται 58 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβεστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 85. I close the vote. Ένας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της mm. έκθεσης. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα, πέρας ψηφοφορίας. «48 προς 1. Συγχαρητήρια στον κύριο Σιγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες μας στην Επιτροπή Ήτρε. Και τώρα ας περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, dear friends, we start with our agenda. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξή μας. Ε, λοιπόν, εξέταση των εκτελεστικών νομοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά ε, τις, ε, τα τέλη σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής και τον σχετική, τη σχετική εκτελεστική πράξη της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, συνάδελφοι. της υπηρεσίας περιαγωγής στο πλαίσιο του κανονισμού για την νέα αγορά τηλεπικοινωνιών, τον κανονισμό TSM, όπως γνωρίζετε, έχουμε και εδώ μαζί μας την συγκήτρια. Ε, σε σχέση λοιπόν με αυτό το κανονισμό υιοθετήσαμε μια γνωμοδότηση, καθώς τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής θα καταργηθούν από τις 15-2017 στο πλαίσιο ενός συστήματος που λέγεται Rome Like at Home, δηλαδή περιαγωγή με κόστος εσωτερικού, με χρέωση εσωτερικού. Ε, και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας η Επιτροπή αποφάσισε ε, ζητήθηκε από εκείνη να υιοθετήσει κάποιους λεπτομερούς ε, κανόνες ώστε ε, να υπάρχει, να προβλεφθεί μια θεμητή χρήση αυτής της υπηρεσίας επενεργογής για να μην γίνει κατάχρηση του συστήματος. Στις 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν η Επιτροπή δημοσίευσε ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης αλλά μετά από κριτική που δέχθηκε και μάλιστα και από την πλευρά του Κοινοβουλίου που είναι πολύ σημαντικό απέσυρε αυτό το σχέδιο, αυτή την αρχική πρόταση και η Επιτροπή σήμερα απέστειλε ένα νέο σχέδιο 15.2.3 το οποίο στις 3 παρατέταρτο συγγνώμη απεστάλλει ε, έχουμε μάλλον ε, στη διάθεσή μας ε, γι' αυτό δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να εξετάσουμε αυτό το σημείο ο Γιώργος Ροπέντο Βιόλα, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διευθυντής Connect, τον καλωσορίζουμε και του δίνουμε το λόγο, είναι δίπλα μου, συγγνώμη. Mr. Chairman. So, first of all, let me... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω λίγο το τι θα πρέπει να κάνουμε για να εφαρμοστεί να εφαρμοστούν οι διατάξει μέσω τη εκτελεστική πράξη. Το σχέδιο λοιπόν το οποίο αποστήλαμε σήμερα στο Συμβούλιο και στην ε, Κοινοβούλιο ε, ε, έχει λάβει τη γνωμοδότηση, ή μάλλον θα λάβει τη γνωμοδότηση τη Μπέρεκ έω τι 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Η Μπέρεκ είναι η Ομοσπονδία των Ρυθμιστικών Αρχών. Και από εκεί και μετά, μετά από αυτή τη γνωμοδότηση 15 Οκτωβρίου, τα κράτη-μέλη θα εξετάζουν αυτό το σχέδιο και στις 23 Νοεμβρίου θα ψηφίσουν επί του σχεδίου. Η Επιτροπή λοιπόν προβλέπεται να υιοθετήσει έως τις 15 ε, Δεκεμβρίου την οριστική Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιε εβδομάδε ακόμα στη διάθεσή μα και το θέλαμε αυτό, δηλαδή να έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα για να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με ε, τα θεσμικά όργανα και την ΠΕΡΕΚ, ώστε να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Και ε, στο πλαίσιο τη ψηφιακή διάκεψη στην Πρατισλάβα θα λάβει χώρα ένα workshop με του ενδιαφερόμενου φορεί σε ό,τι αφορά ακριβώ την εκτελεστική πράξη, σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα τέλη περιαγωγή. Αυτή η εκτελεστική πράξη τρέχει ε, ταυτόχρονα με τον κανονισμό για τι ε, αγορέ χοντρική, την περιαγωγή χοντρική, ο οποίο εξετάζεται από κοινού βέβαια από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασία ε, συναπόφαση και ο οποίο πρόκειται να εγκριθεί ω τα τέλη του έτου έξι μήνες δίνονται με αυτόν τον τρόπο στους, ε, ε, στις αγορές ε, παροχής των σχετικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη το νέο σύστημα έως τον Ιούνιο του 2017. Όπως γνωρίζετε, πράγματι αναθεωρήσαμε το σχέδιο που υποβάλαμε με βάση τα όσα μας είπαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς αλλά και το Κοινοβούλιο δηλαδή και την κριτική που μας ασκήθηκε και η νέα τώρα εκτελεστική πράξη, το νέο σχέδιο εκτελεστική πράξη ε, προβλέπεται να είναι πιο σαφή, πιο ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την τήρηση αυτή τη αρχή του Rome like at home, ε, δηλαδή περιαγωγή με χρέο εσωτερικού. Και όπω προβλέπει και ο κανονισμός, ε, αυτό το κόνσεπτ, αυτό, το σκεπτικό σκοπεύει στο να δίνει τι ίδιε τιμές στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιαγωγή του όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρόκειται για ε, κάτι πολύ ε, απλό, δηλαδή ο απλός πολίτης όταν θα ταξιδεύει στην Αλλοδαπή δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα, αυτομάτως θα ενεργοποιείται ακριβώς η μη χρέωση, αν θέλετε, στην περιαγωγή. Ε, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνονται κάποιες, κάποιοι έλεγχοι για παράδειγμα, ε, εάν υπάρχουν κάποιες κάρτες SIM ε, στις οποίες δεν υπάρχει κάποια χρήση τους, καμινερνική χρήση ή όταν, για παράδειγμα, ε, γίνεται χρήση μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα πουθενά αλλού ή όταν έχουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση ενός ατόμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος για μία σειρά από διαφορετικές SIM. Και επίσης έχουμε δώσει τη δυνατότητα στις μυστικές αρχές να κάνουν ελέγχους σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος ο οποίος μεταπολεί κάρτες SIM. Ε, το σύστημα λοιπόν ε, είναι πολύ απλό για όλους τους μη μπλεκόμενους άμεσα στη διαδικασία, δηλαδή απλώς θα ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτή roam like at home χωρίς δηλαδή επιπρόσθετη χρέωση ε, και αυτό βέβαια είναι αντίστοιχο με, το, τα όσα ισχύουν και σε ό,τι αφορά και το επίπεδο της χοντρικής που έχει συζητηθεί τώρα. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων που θα διαξάγουν οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα είναι αρμόδιες και για την εποπτεία της στήριξη των κανόνων, θα έχουν λόγω αρχέ και ε, την αρμοδιότητα για να λαμβάνουν αποφάσει όταν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι εξαιρετικέ ε, περιπτώσεις. Καταρχήν ω προ υπάρχουν και από εκεί και μετά, εάν για παράδειγμα πρόκειται για ε, περίπτωση μεταπόληση, θα μπορεί να προβαίνει σε μπλοκάρισμα, σε φραγμό των σχετικών καρτών, αλλά θα πρέπει να προβαίνει και σε μια σχετική ενημέρωση της ΕΜΑΡΗ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, αλλά βέβαια επειδή πρόκειται και για το μακέτο βιωσιμότητα στο sustainability pact το οποίο αφορά ο κανονισμός, θα δώσω το ρόγο αν μου επιτρέπετε στο συνάδελφο. Πρόεδρος, ε, ναι, κύριε Γενική Διευθυντά, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στους ε, πολίτες μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ και τον Διευθυντή Άντωνη Γουίλαν, για μια πολύ σύντομη παρέμβαση, γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο κατάλογο μελετών. Οπότε ίσως καλύτερο θα ήταν να ε, μη σπαταλήσατε πολύ χρόνο τώρα, ούτως ώστε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην απάντηση των ερωτημάτων που θα θέτουν οι συνάδελφοι. Γιατί άλλωστε οι συνάδελφοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το, το ζήτημα, γιατί το ίδιο έχουμε εξετάσει από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ε, ε, ε είναι προσθήκη στα όσα είπε ο συνάδελφος. Ε, να πω ότι υπάρχει και ένας ακόμα πυλώνας που θα πρέπει να θετήσουμε στις 15 Δεκεμβρίου σε επίπεδο εκτελεστικό δηλαδή ε, σε ό,τι αφορά τις παρεκκλήσεις ε, βιωσιμότητας sustainability, ε, για το sustainability και αυτό αφορά περιπτώσεις όπου εάν εφάρμοζε με αυτόν τον τρόπο ο πάροχος των υπηρεσιών το σύστημα οι, υπηρεσίες του ουσιαστικά θα ήταν υποκίνδυνο. Δηλαδή ουσιαστικά για περιπτώσεις όπου ε, θα δημιουργούνταν αυτό το φαινόμενο όπως λέγεται το waterbed όπου ουσιαστικά θα οδηγούσε σε αύξηση των, ε, ε, των τιμών στην εσωτερική αγορά του εν λόγω κράτους μέλους. Άρα λοιπόν στο σχέδιο εκτελεστικής πράξης που σας υποβάλλουμε αναφέρεται το όριο του 5% για δυνητική μείωση των πωλήσεων σε επίπεδο λιανικών ε, πωλήσεων για το συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών, ούτω ώστε κάτι τέτοιο να δικαιολογεί, δηλαδή το 5% μια πιο προσεκτική εξέταση από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, αλλά από εκεί και μετά. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η, μπορεί, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να ε, αρνηθεί ε, την, την παροχή αυτής της εξαίρεσης σε περίπτωση για παράδειγμα προστασία συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών ή σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να συμβεί, δηλαδή η μείωση των πωλήσεων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συζητητές, αλλά ε, σας παρακαλώ όλοι σας να περιορίσετε το χρόνο της αγόρευσή σας σε 1,5 λεπτό. 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Πολύ σύντομα ερωτήματα να θέσετε λοιπόν. Ε, κυρία Δικαστήλο, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο μιλητές, και τον κύριο Βιόλα και τον κύριο Βίλαν. Κοιτάξτε, μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, και λέω αποτυχημένη όχι γιατί δεν μπόρεσε να καλύψει τους στόχους, αλλά γιατί δημιουργήθηκε τεράστια σύγχυση από τα τις 90 ημέρες που είχαν προταθεί. Βρισκόμαστε τώρα ενώπιον σε μια, μιας πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λύνει όλα τα προηγούμενα ε, ε, προβλήματα εγγυάται το Rome like at home, ότι η περιεγωγή θα είναι σαν να είσαι στην πατρίδα σου. Ε, διασκεδάστηκαν διάφορες αμφιβολίες και φόβοι και αυτά έχουν να κάνουν με την εποπτεία ακριβώς αυτής της ρήτρα ε, της λελογισμένης ε, χρήσης. Είχα την ευκαιρία πολύ γρήγορα να διατρέξω το κείμενο γιατί ήρθε η τελευταία στιγμή. Θα επιθυμούσα να ληφθεί υπόψη να υπάρχει κάποια δυνατότητα ένας μηχανισμός ούτως ώστε εάν παρατηρηθεί καταχρηστική ε, συμπεριφορά από δεσπόζουσα θέση του παρόχου αυτό να κοινοποιείται και να μπορεί να απαντήσει ο συνδρομητής, εκείνος που έχει δηλαδή το, το πακέτο με την εταιρεία πριν ε, του επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο ή ε, έξοδα ε, επιπλέον. να ειδοποιείται δηλαδή ο συνδρομητής έτσι ώστε να ε, είναι οι καταναλωτές πιο ήσυχοι και να ξέρουν ε, να κανονίσουν την πορεία τους. Κατά τα άλλα τα βλέπω και τα θεωρώ όλα αυτά πάρα πολύ λόγικα και συμφωνώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ ήταν η, κυρία Δελκαστήγιο, η κυρία Τόγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σύμφωνα με τα όσα μόλις υπόθηκαν ως εκτίμηση για αυτή τη θέση που πιστεύω ότι συγκεντρώνει όλα τα σημεία, συντονίζει τα πάντα, δηλαδή το να διατηρήσουμε την νομοθετική μας δέσμευση για άρση των χρέωσεων περιαγωγής, αλλά και να έχουμε και μια δίκαιη χρήση. Δηλαδή όλα αυτά να γίνουν με λογικό, σωστό τρόπο, χωρίς παραθυρακία για καταχρήσεις. Τώρα, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω και φυσικά θα εμβαθύνουμε στο μέλλον, αλλά θέλω να δούμε αυτή την προσέγγιση. Υπογραμμίζω λοιπόν το εξή. Πρέπει, όπως είπε ο κύριος Βιόλα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς υποχρεώσεις για το χρήστη, αλλά αν και αυτός ο χρήστης αντιληφθεί ότι δεν, ε, αν δεν έχει χρεώσεις που βρίσκεται, που ζει, δεν πρέπει να αναφέρει που ταξιδεύει κτλ. Αλλά σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια ύποπτη κίνηση ε, στο δικό του φάκελο να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να μπορεί να καταλήξει σε μπλοκάρισμα της κατάκρισης αλλά όχι να ελέγχουμε τις δραστηριότητες του καθενός δηλαδή αυτό το σύστημα προειδοποίηση όπως είπε η Πιλάρ και η επαλήθευση και εγώ θα έλεγα οι δημόσιες αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές ε, να μην ε, αναθέσουν στους φορείς κάποιο καθήκον που δεν είναι δικό τους αλλά φυσικά ναι, έχουμε και την οικονομική λογική που ε, επιβάλλει κάποια ανώτατα όρια, ελπίζω να είναι λογικά, να έχουν υπολογιστεί σωστά ε, και προ όφελο των φορέων, αλλά ξέρετε μερικές φορές και ε, ο φορέας χρησιμοποιεί κανόνες για να φταίνουν τα κέρδη του, δηλαδή πρέπει και αυτοί λογικά να θέτουν τα ανώτατα όρια. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ε, ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκτιμώ αυτή την προσπάθεια ευρεία συζήτησης ε, για αυτή την περίπλοκη πρόταση για την περιαγωγή. Μια περίπλοκη βλέπω εγώ. Ε, κάποιοι όροι ορολογίας, κάποιες πτυχές που ανέφεραν μόλις συνάδελφοι, δημιουργούν ε, πρόβλημα και ελπίζω να το διευκρινίσουμε με την ΠΕΡΕΚ για παράδειγμα όταν μιλάμε για παράδειγμα για μεγάλες περιόδους αδράνειας όπου θα πραγματοποιούνται και ποια έλεγχη δεν είναι απολύτως σαφές πιστεύω κοιτώντα το κείμενο βάσει των συζητήσεων μας ε, ελπίζω με την ΠΕΡΕΚ και με τους επιμέρους φορείς να μπορέσουμε να την απλοποιήσουμε διότι προφανώς ε, δεν έχουμε προλάβει να το μελετήσουμε λεπτομερώς, αλλά μου φαίνεται πολύ περίπλοκο. Και έτσι η επίβλεψη και ο έλεγχος θα περιπλέκονται, οπότε ελπίζω να ε, η συζήτηση που κάνουμε τώρα να είναι μόνο η αφετηρία. Παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο ε, πριν τα δελτία του Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ κύριε συνάδελφε, κυρία Κάλλας εκ μέρους του Αλντε. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μας ομάδα καλωσορίζει την αναθεωρημένη πρόταση. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, οπότε δύο ερωτήσεις μόνο για την ε, εκτελεστική πράξη στις αιτιολογικές σκέψεις. Αναφέρεται ότι θα ζητείτε το κράτος ε, ε, κατοικίας ε, για την ε, περίπτωση κατάχρησης, δηλαδή μόνο σε περίπτωση κατάχρηση θα ζητείτε ποια είναι η κατοικία του πελάτη. Οπότε ρωτάω ουσιαστικά το αίτημα για ε, έγγραφα που να αποδεικνύουν την κατοικία του πελάτη είναι κάτι που προβλήθηκε μόνο για αυτές τις περιπτώσεις το ρωτάω διότι και για τις προπληρωμένες κάρτες αν είναι να παρέχονται τέτοια έγγραφα αυτό μπορεί να αυξήσει το φόρτο εργασίας. Τώρα όσον αφορά την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων ο φορέα τη περιαγωγή μπορεί να εφαρμόσει αναλογικούς μηχανισμούς για να αποφύγει την κατάχρηση της περιαγωγή. αλλά αφού δεν υπάρχει περιορισμός σε ημέρες, κάτι καλό φυσικά πιστεύω, έχει αφαιρεθεί ο αριθμό, αλλά δεν υπάρχει και περιορισμός ε, του διαστήματος ε, για το οποίο θα διατηρεί τα στοιχεία του καταναλωτή ο φορέας. Μπορεί να το αναλύσει λίγο η Κομισιόν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλάς ο κύριος Ρέμον εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Με την ε, πρόταση συμφωνώ ότι μπορούμε να εργαστούμε. Ε, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τις ημέρες τώρα. Πόσες μέρες το αφήνουμε στην αγορά με επιβάση... Ε, ε Ποιο στοιχείο μπορείτε να θεωρήσετε ότι θα είναι λιγότερο από 90 ημέρες και ποιο το ορίζει αυτό η διατησία και πώς βεβαιώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι καλύτερο ε, αυτό για τους καταναλωτές από τις 90 δωρεάν ημέρες. Έχετε στοιχεία αυτό για να το τεκμηριώσετε έρευνα και αν υπάρχει πραγματικά ε, σκληρός ανταγωνισμός για τη λελογισμένη χρήση, πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα επιβιώσουν, δεν θα επιβλέψουν ένα σε δύο πάροχοι ένα χώρα που είναι παρόντες εις βάρος των μικρών. Δεν τα έχω καταλάβει αυτά πάρα πολύ καλά. Μπορούσατε να με διαφωτίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορέλη, από την Ευθυντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είδα την πρόταση πριν από μια ώρα, οπότε με μια πρώτη ανάγνωση εντόψα τρία προβλήματα. Πρώτον, σύμβαση μεταξύ πελάτη και φορέα. Δεν μπορεί να είναι δεσμευτική μόνο για τον πελάτη. Η Κομισιόν λοιπόν πώς προβλέπει να αποφύγει ο φορέας να έχει τα κινητρά, να διακινδυνεύσει τα δικά του κέρδη ε, κατά, ε, προς ε, ε, δημιουργώντας ζημιά στον καταναλωτή σε περίπτωση που διότι δεν είναι βιώσιμη δηλαδή το πρόγραμμά του μπορεί να ζητήσει αύξηση της τιμολόγησης του roaming. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι θα γίνονται επαληθεύσεις για αποφυγή των καταχρήσεων ή κομισιών πώς σκοπεύει να αποφύγει να παρέχει τεράστιες δυνατότητες απόφασης στους φορείς. Και μετά υπάρχει το θέμα της του χρονοδιαγράμματος το Δεκέμβριο που θα υιοθετηθεί η νέα εκτελεστική πράξη με τα ανώτατα, τα όρια των ε, τιμών περιοχής. Δεν θα έχουν ακόμα οριστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καπέλ, εκ μέρους του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιχαίρω την υποβολή αυτού του νέου ε, σχεδίου γιατί πραγματικά έχει διαμορφωθεί πολύ θετικά μετά από την τελευταία ε, συζήτηση ε, που κάνουμε και μετά από την ε, συνάντηση που είχαμε στις 13 Σεπτεμβρίου και με τον Επίτροπο Έττιγεν και τότε βέβαια η εν λόγω πρόταση προέβλεπε μόνο 90 μέρες. Πραγματικά έχει γίνει σημαντική πρόεδρος, πρόοδος συγγνώμη, σε αυτό το νέο σχέδιο και έχει πραγματικά κινηθεί ταχύτατα εδώ η Επιτροπή τους ώστε να πάυσει να υπάρχει αυτό το όριο των 90 ημερών που επιβάρυνε τον καταναλωτή και να προσπαθήσουμε τελικά να επιτύχουμε τον ε, στόχο που είμαστε θέσει ευθύ εξ αρχή, δηλαδή την κατάργηση των ε, τελών επιρρεγωγή έω τον Ιούνιο. Τώρα τέθηκε και είχε τεθεί και στο πλαίσιο του διαλόγου με τον κύριο Ότιγκεν αυτό το ερώτημα, δηλαδή του πώ θα γίνεται η διαπίστωση τη κατάχρηση και πώ θα ορίζεται αυτό. Ε, νομίζω λοιπόν που σχετική ε, συνάντηση που θα γίνει και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί οι ρυθμιστικές αρχές τώρα θα έχουν μία σειρά από νέες ευθύνες ώστε να καταπολεμούν την κατάχρηση και προκειμένου να συλλέγουν τα ε, σχετικά δεδομένα. Οπότε τίθεται το ερώτημα θα έχουν τους κατάλληλους πόρους αυτές οι αρμόδιες αρχές στη διάθεσή τους για να το κάνουν και ε, ποια θα είναι τα στοιχεία που θα τους επιτρέπουν να εντοπίζουν την κατάχρηση. Οπότε ε, θα ήθελα, ε, περιμένουν αυτές οι Πάντω Πάντως ε, θεωρώ πολύ ε, σημαντικό στο νέο σχέδιο ότι δεν ισχύει πάντα αυτό το όριο των 90 ημερών. Και από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα των, του ερωτήματος του πώ γίνεται η, ο υπολογισμό των διαφόρων τελών ή μη τελών όταν ο πολίτης δεν ταξιδεύει μόνο σε ένα αλλά σε πολλαπλά κρατημέλη γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βέβαια το κάνουν αυτό συχνά. Η κυρία γιατι υπαρχουν καποιοι οποιοι βεβαια το κανουν αυτο συχνα η κυρια Φόρτζ. Φόρτ, συγγνώμη, ε, ε, η πρόεδρος της Επιτροπής ΕΜΚΟ και παίρνει τον ε, λόγο στα πλαίσια του άρθρου 54. Ε, πράγματι, Πρόεδρε, με ενδιαφέρει από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες προστασίας του καταναλωτή. υποστηρίζω πλήρως την προσέγγιση του Room Like at Home της περιαγωγής δηλαδή με χρέος εσωτερικού, αλλά ε, ανησυχώ ότι δεν είναι η εν λόγω πρόταση αρκούντος σαφής και κατά συνέπεια θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική εφαρμογή της από τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Ε, ε, στις προτάσεις τις οποίες διαπραγματευτήκαμε είχε καταστήσει σαφές ότι η θεμητή αυτή χρήση, η χρήση το Φέργιους προβλέπεται για περιοδική ε, για περιοδικά ταξίδια οι μεταβάσεις ε, στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν προβλέπω να παρέχει πρόσβαση εάν δεν πρόκειται για ε, περιοδικά ταξίδια. Για να σας να δώσω το παράδειγμα. Δεν θα να παίρνει κανείς ε, μία πτήση της Ryanair και να, παραμένει, να περιμένει συγγνώμη, από την British Airways να ε, παράσχει την ίδια τιμή για να, ε, πρώτη θέση. ουσιαστικά με αυτή την πρόταση που κάνει με την στρατηγική για τη θεμητή χρήση κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή ουσιαστικά εστιάζει μόνο στην κατάχρηση ό,τι αφορά αυτή την θεμητή χρήση. Και ναι, προφανώς θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι οι, ε, ε, οι που έχουν λιγότερες δαπάνες εδώ δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τους καταναλωτές με υψηλότερες δαπάνες. Και από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κινούνται διασυνοριακά. Αν είναι κανείς δηλαδή ε, φοιτητή, για παράδειγμα, θα είναι πολύ δύσκολο να ε, αποδείξει, να τεκμηριώσει ότι υπάρχει πραγματικά αυτό το περιοδικό ταξίδι. Ίσως να υπάρξει πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει μία ε, πτυχή την οποία θα έπρεπε να είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τακτικότητα των ταξιδιών, σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα τα λάβει αυτά υπόψη στο σχέδιο τη εκτελεστική πράξη. Διαφορετική περίπτωση φοβούμαστε ότι η Επιτροπή δεν θα τηρήσει τα πλαίσια τη εντολή που έχει λάβει. Ε, θα ήθελα ένα λεπτό υπολοιπτό συνάδελφε να αγοράσω. Παρακαλώ. Συνάδελφο Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον ε, πρόεδρο Γιούνκερ, ο οποίο βέβαια έδωσε το έναυσμα για να υποβληθεί το νέο σχέδιο. Και αυτό γιατί, για να είναι σαφέ για τον καταναλωτή ότι όταν ε, προβαίνει στη σύναψη ενό ε, συμβολέου, στην πατρίδα του θα μπορεί να χρησιμοποιεί την ελόγω σύνδεση με τον ίδιο τρόπο και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζουμε ότι και αλλού υπάρχουν όροι κατάχρησης όλων των παρόχων αυτών των σχετικών υπηρεσιών. Στα συμβόλαια δηλαδή προβλέπεται κάτι τέτοιο, προβλέπονται δηλαδή περιπτώσεις κατάχρησης ε, και στο πλαίσιο δηλαδή του συμβολέου στην, ε, στην αγορά του κρατούς μέλους. Από εκεί και μετά ε, υπάρχουν δηλαδή περιπτώσει όπου υπάρχουν διαφορέ τη τάξη του δεκαπλασίου και ε, ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη, οπότε θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και μέσα στα τρία χρόνια που μα, αποβαίνουν, δηλαδή έω το 2019, θα πρέπει να έχουμε εφαρμόσει τον, ε, με τέτοιο τρόπο την περιαγωγή το Rome like at home, ούτως ώστε να έχει πράγματι εφαρμοστεί στην πράξη η νέα αγορά τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Κουπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θεωρώ πως ε, πρόκειται ε, εδώ για ένα ε, θετικό βήμα προκειμένου να ε, διασφαλίσουμε το, να μην δενιστούν τελικά οι αγορές λιανικής περιαγωγής για να φτάσουμε στον στόχο που θέλαμε και νομίζω πως αυτό ευθυγραμμίζεται και με τη σχετική έκθεση που προετοιμάζουμε. Δηλαδή, εάν σε, σε επίπεδο της χοντρικής δεν υπάρχει επιπρόσθεση χρέωση, τότε δεν θα χρειάζεται να προβλέπουμε και διάταξη σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα. Γιατί είναι πολύ άσχημο το να λέμε ότι μια νομοθεσία είναι διαμορφωμένη με αυτόν τον τρόπο, ούτω ώστε να υπάρχει ο κίνδυνο κάποιοι από του παίκτε στην αγορά να ουσιαστικά να μην μπορούσαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του. Και είναι συνδεδεμένο προφανώ με αυτόν τον κανονισμό, γιατί αναφέρεται εδώ στο άρθρο 5 τη πρότασή σα ότι εάν ο πελάτη πράγματι καλείται να ναι. Ε, καταβάλει μια χρέωση, τότε αυτή ε, αποτελεί τμήμα τη ε, χρέωση σε επίπεδο χονδρική, όπω είχαμε προβλέψει. Τώρα να θέσω κάποια ερωτήματα, δύο ερωτήματα διασφαλίζεται ότι αυτή η διάταξη δεν αποτελεί ουσιαστικά ένα παραθυράκι στον νόμο, ώστε ο, ε, ε, ο πάροχο των υπηρεσιών ε, να μην καλείται να καταβάλει τίποτα για την περιαγωγή. Και μετά, δεύτερο, πώς θα διαπιστώνουμε αν κάποιος χρησιμοποιεί ε, περισσότερε από μία Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή που αντέδρασε ε, στις, στην κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απέσυρε την προηγούμενη πρόταση για να επιβάλλει μια νέα πρόταση την οποία θεωρούμε πως είναι πολύ καλή, πολύ καλά οργανωμένη ε, και για μας βέβαια το ζήτημα της περιεχογής και της ελεύθερης Ευρώπης ε, μας απασχολεί εδώ και 25 χρόνια και για μας είναι σημαντικό να τηρήσουμε την πολιτικού χαρακτήρα υπόσχεση που δώσαμε ε, στους πολίτες μας ότι δηλαδή το room like at home, η περιεγωγή όπως το σπίτι να εφαρμοστεί πράγματι στην πράξη. Πρόκειται δηλαδή για μια κλασική περίπτωση που θα πρέπει να προβλέψουμε σαφείς κανόνες. Θα πρέπει δηλαδή ε, ρυθμιστικά να προβλέψουμε μια λύση η οποία θα αποτρέπει την κατάχρηση και θα ήθελα να ε, ρωτήσω εδώ, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει ε, υποψία κατάχρησης, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παύσης του συμβολέου, ακύρωση του συμβολέου, αλλά να υπάρχει μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία να επιτρέπει το αν κατά πόσο έχει λάβει η χώρα κατάχρηση ή όχι. Πάντως, με πολύ λίγες εξαιρέσεις ο δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε βέβαια αυτή την λύση που θέλαμε και να έχουμε τη λύση την επίσης υπόσχεση που είχαμε δώσει στους πολίτες μας για το Ρώμουλα Κατοχό. Ευχαριστώ. Όταν ε, εγκρίναμε το TCM εγώ ψήφισα ε, και το Κοινοβούλιο να καταργηθεί το roaming. Ε, σήμερα μας έρχεται η δεύτερη πρόταση, δεν μπόρεσα να αφήνω. η πρώτη δεν ήταν καλή. Τώρα η μουσική ωραία ακούγεται, αλλά για να δούμε πώς θα ε, εφαρμόσουμε στην πράξη. Δεν θα πρέπει να γίνει πεδίο εχθροπραξιών η σχέση ε, καταναλωτή με πάροχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ε, τα πράγματα στα χέρια των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων της αγοράς θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκληθούν τώρα αυξήσεις στα τιμολόγια ε, των ε, καταναλωτών των χωρών που υποδέχονται εκείνους που έχουν το roaming. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω. Ε, καλωσορίζω την πρόταση αυτή για ένα μοντέλο που έρχεται να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις ε, σχετικές με τη βιωσιμότητα του μοντέλου της περιαγωγής, το περίφημο Rome Like at Home. Αν θέλουμε όσο γίνεται περισσότεροι να υποφελούνται αυτού του συστήματος που το επιθυμούμε και το καλωσορίζουμε πρέπει να κατανοήσουμε ότι και οι πάροχοι και οι εταιρείε θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλιώς θα έχουμε υπερβολικές χρεώσεις. Και σας ερωτώ πώς ε, προτίθεστε εσείς να εγγυηθείτε ε, αυτό το γεγονός ότι ουδής πρόκειται να ξεπεράσει αυτά που λέει ε, η ε, πρόταση και η απόφαση. Μπορεί να είναι καλόπιστοι οι καταναλωτές και καλόπιστοι κάποιοι πάροχοι, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι κακόπιστοι. Τι θα γίνει εκεί, η κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση, Rome Like at Home, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, γνωρίζουμε ότι οι πολίτες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Εγώ είμαι Φιλανδή και στη Φιλανδία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για δεδομένα και είναι πολύ φθηνά. Ε, και τώρα θα είναι μεγάλη ε, η επιβάρυνση για τους παρόχους στη Φιλανδία αν είναι δωρεάν ή χρήση αυτή. Τι γίνεται λοιπόν με τα δεδομένα. Αν δεν υπάρχει ένας μέσος όρος ή αν μπορεί ο κάθε καταναλωτής απεριόριστα να κατεβάσει περιεχόμενο, τι θα γίνει. Δεν θα επιβαρυνθούν ε, οι εταιρείε υπερβολικά. Δεν προτείνεται να προτείνετε όρια. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πράγματι ε, μια πολύ σημαντική ε, πρόταση αποτέλεσμα αφημιβασμού και προφανώς πολύ σημαντική για τους πολίτες μας. Τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι να υπάρξει ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο σε εθνικό πλαίσιο και υπάρχει βέβαια και η πρόκληση της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα, δηλαδή να λάβουμε το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο είναι σημαντικό για την οικονομία μας και όταν θα περάσουμε στη φάση της αξιολόγησης, θα πρέπει να ε, διαπιστώσουμε ότι έχει ε, θετικό αντίκτυπο τόσο στους πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν, όσο και για τους παρόχους των υπηρεσιών. Ε, και αυτό βέβαια και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε γενικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Ο Επίτροπος ο κ. Κανιέτε είναι καθοδόν, αλλά έχουμε ακόμα πέντε λεπτά για να Απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Το συντομότερο δυνατόν και όσο πιο εύστοχα γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλες αυτές οι ερωτήσεις ε, χρήζουν απάντησης. Θα στείλουμε ε, τις μεγάλες απαντήσεις ε, γραπτός στη γραμματεία σας. Τώρα θα δώσω κάποιες σύντομες απαντήσεις προς το παρόν. Ε, για τις οι πρώτε ερωτήσει από την κυρία Καστίγιο και την κυρία Τόγια είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τη ρυθμιστική αρχή και του πελάτη. Να το πω πολύ γρήγορα τώρα και για να απαντήσω και στην κυρία Νίπελ. Το σύστημα είναι προοδευτικό για τον πελάτη. Ο κανονικό πελάτη δεν έχει κάτι να κάνει. Υπάρχει μια συνδρομή, ένα κανονικό συμβόλαιο, οπότε το Home δίνεται στο πλαίσιο αυτού. Τώρα, σε περίπτωση που κάτι παράξενο συμβεί, για παράδειγμα ε, μετακόμιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα, θα λάβει ένα SMS. Δηλαδή συνεχίζει το Roam Like at Home και μετά αυτός ο πελάτης μπορεί να διαμαρτυρηθεί στον φορέα. Αν ο φορέας δεν απαντήσει, ενώ υποχρεούται να απαντήσει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στη ρυθμιστική αρχή για να διευθετήσει την υπόθεση. Οπότε δεν θα αποσυνδεθεί ο πελάτης, δεν θα διακοπεί η σύνδεσή του, απλά θα λάβει μια ειδοποίηση ότι το σύστημα έχει ανεχνεύσει ε, μη φυσιολογική χρήση του Rome Like at Home. Αλλά δεν πρόκειται να διακοπεί η σύνδεσή του. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όπου ο ανακαλύπτει μια οργανωμένη ε, επιχείρηση ουσιαστικά παράνομη, μια, οργανωμένες συναλλαγές παράνομες όπου πολλές ε, κάρτες ε, πολλούνται στο εξωτερικό. Αυτές πρέπει να διακοπούν αμέσως, αλλά ο φορέας πρέπει να ενημερωθεί αμέσως φυσικά και η ρυθμιστική αρχή. Και η ρυθμιστική αρχή εκεί έχει να λάβει την τελική απόφαση. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις. Οι μονομένοι πελάτες δεν έχουν να για κάτι. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί, από το σύστημα κάποιο μη φυσιολογικό μοτίβο χρήση θα λάβει ένα SMS χωρί όμω αποσύνδεση ούτε διακοπή τη σύνδεσή του ούτε διακοπή του ROM Black and Home και φυσικά έχει ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στη ρυθμιστική αρχή, στη ρυθμιστική, ρυθμιστική αρχή στον φορέα για να επιλύσει το ζήτημα. Κύριε Τωσανόφσκι, για το μεγάλο χρονικό διάστημα, όπω λέτε και εσεί, πρέπει να συζητήσουμε με την Μπέρεκ για τι λεπτομερεί ρυθμίσει, αλλά επαναλαμβάνω, ένα κανονικό πελάτη ε, δεν θα επηρεαστεί από αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τις ακραίες περιπτώσεις. Ε, ε το αίτημα για έγγραφα, όπως είπα, δεν είναι κάτι που θα συμβαίνει. Κανονικά ο κόσμος έχει μια πιστοτική κάρτα και αυτό αρκεί. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ζητείτε ταυτότητα για μια συνδρομή σε κινητή τηλεφωνία. Σε άλλα κράτη όχι. Τώρα, ειδικότερα στις περιπτώσεις των προπληρωμένων καρτών, φυσικά ένα χρήστη μπορεί να αγοράσει όσε θέλει, σε όποια χώρα θέλει. Αλλά αν θέλει να έχει το Rome like a home ενεργοποιημένο σε μια χώρα, πρέπει να δείξει κάτι για αυτή την προπληρωμένη κάρτα. Δικότερα να έχει χαμηλή πίστοση ότι έχει κάποια σύνδεση με τη χώρα. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω στον κύριο Ρεν. Ρώτησε τι αλλάζει εντό 90 ημερών. Αυτό είναι το θέμα. 90, για το 90-95% των πελατών δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που αλλάζει για παράδειγμα για ένα φοιτητή Εράσμου, ο οποίο θέλει να ενεργοποιήσει το Rome Like at Home σε μια χώρα που δεν έχει καμία δραστηριότητα και η ταυτότητα δεν δείχνει ότι είσαι φοιτητή του Εράσμου. όπου το κανονισμό λέει και τέθηκε και ερώτημα γι' αυτό, Μπορεί να πάει κανείς με την κάρτα Εράσμου οποιοδήποτε αποδεικτικό και να ενεργοποιήσει το Rome Like at Home στη χώρα όπου βρίσκεται για το πρόγραμμα Εράσμου. Αυτή είναι η διαφορά ε, σε σχέση 90 μέρες. 90 μέρες ήταν κάτι πιο αυστηρό εδώ τώρα για κάποιες ε, περιπτώσεις κάπως ακραίες ε, πρέπει ζητείτε να αποδείξει κανείς ότι έχει κάποια σχέση με τη χώρα, δηλαδή ότι είναι προσωρινά εκεί αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα φοιτητής, για παράδειγμα του Εράσμους και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να το ενεργοποιηθεί το Roma Like a Home. Όπως είπα είναι σταδιακά, είναι, λειτουργεί προοδευτικά το σύστημα. Ε, τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου, θα χρειαστεί να την αναθεωρήσουμε αλλά δεν προβλέπουμε μεγάλες διαφορές. Διότι δεν είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις ε, όπου ο οικονομικός αντικτύπωση είναι σημαντικός. Για να απαντήσω και στην κυρία Φόρντ εδώ, έχουμε εξετάσει προσεκτικά όλα τα μοτίβα των ταξιδιωτών και των συνηθιών ταξιδιού στην Ευρώπη. Έχουμε πολλά στοιχεία ώστε να είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμο το σύστημα. Κύριε Μπορέλη, τώρα η διακριτική ευκαιρία του φορέα θα περιορίζεται, όπως είπα, από το σύστημα ελέγχων, αστηρών ελέγχων από τη ρυθμιστική αρχή. Οι ελευθερίες δηλαδή που θα έχει να δράσει ο φορέας. Ναι, πράγματι κύριε Κάβελ, θα χρειαστεί να συζητήσουμε λεπτομερώς με την Μπέρεκ τις λεπτομέρειες όσον αφορά την γλώσσα και την αλληλεπίδραση και την ορολογία μεταξύ ε, ε, φορέα και ρυθμιστικής αρχής και πελατών. Και με βέβαιο ότι η Μπέρκ θα κάνει κάποιες πολύ εύστοχες προτάσεις. Τώρα, για κάποια ζητήματα ανέφερε και κ. Νίκα την ε, βιωσιμότητα. Επαναλαμβάνω. Και σε αυτή την περίπτωση. Ας δούμε και έτσι απαντώ και στην κυρία Καπουλανάτρη. Ας δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του συνομοθέτη. Και φυσικά θα υπάρχει ε, ε, κάποια σύνδεση μεταξύ του συστήματο αυτού και των ε, κανονικών τιμών. Κύριε Βυρκούνεν, πράγματι, η ιδιαιτερότητα των χωρών του Βορρά πρέπει να ξαναμελετηθεί με την Μπέρεκ. Αναφέρομαι τώρα δηλαδή στα ε, προγράμματα περιόρισης της δεδομένων που δεν ε, συνηθίζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να συζητηθεί με την ΠΕΡΕ και θα επανέλθουμε όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις. Ε, σε περίπτωση ε, του cross-subsidy της διασταυρούμενης ε, επιδότησης ελπίζω ότι εδώ έχουμε αποφύγει αυτή την, ε, αυτό τον κίνδυνο γιατί αυτό σχετίζεται με τον πελάτη. Και αυτό θα είναι σημαντικό και θα το συζητήσουμε με την Πέρα, κύριε Ρούμπιχ. Όπως είπαμε, είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες που έχουν μια φυσικολογική συνδρομή να λαμβάνουν το Roam Like at Home και οι άλλοι πελάτες θα ε, πρέπει να πάρουν κάποια στοιχεία. Ωραία, ευχαριστούμε πολλά κύριε Γενική Διευθυντή. Αγαπητοί συναδελφοί, είμαι βέβαιος ότι όλες σας οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές για την κοινή γνώμη. Όλα ό,τι συζητάμε τώρα θα μεταδοθεί live στο διαδίκτυο. Έχουμε λοιπόν στα χρήμα μας τις ερωτήσεις. Να σας ζητήσω κύριε Γενική Διευθύντα ε, και ευχαριστώ ξανά για την παρουσία σας εδώ. Απαντήστε τις ερωτήσεις γραπτός. Εμείς θα τις πάρουμε, θα τις στείλουμε στα μέλη μας, ώστε να λάβετε τις απαντήσεις, τις λεπτομερείς απαντήσεις για τις ερωτήσεις σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι πολίτες μας θέλουν να έχουν πλήρη ενημέρωση. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή χρόνο για να ε, μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε ο Επίτροπος ο κ. Κάνια να περιμένει μπροστά στην πόρτα, γιατί μαζί μας είναι, με το μέρος μας είναι, απλά πίσω από την πόρτα. Ε, οπότε θα σταματήσουμε τώρα και θα λάβετε εσείς τις απαντήσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε γραπτή μορφή και μετά θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αν δεν συμφωνείτε ή θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, μπορούμε να τα ξαναστείλουμε όλα αυτά ως ερωτήσεις επιπλέον παρατηρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σημαντική διαδικασία. Μια τελευταία ερώτηση τώρα. Πότε να αναμένουμε τις απαντήσεις σας, κύριε Γενική Διευθυντή. Όπως είπα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακούσαμε σήμερα και τον κυριο βελλαν Γουέλλαν φαντάζομαι δύο-τρεις μέρες. Δύο-τρεις μέρες είναι δυνατόν να σας στείλουμε λεπτομερείς απαντήσει οι οποίε θα επικαιροποιηθούν όταν θα έχουμε και τι άλλε απαντήσεις. Μέσα στα τέλη τη εβδομάδα δηλαδή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και να καλωσορίσω τον Επιτρόπο Μιγκελαρία Αρίας Κανιέτε. Ζητώντας του συγγνώμη που σα ε, κρατήσαμε να περιμένετε, αλλά η περιαγωγή είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το ίδιο σημαντική όπως και το ίτερ. Όχι ίτρε, το ίτερ. Uh, uh, σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Περνάμε αμέσω στο επόμενο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ορισμένοι από εμά ενδιαφερόμαστε σφόδρα. Έχει να κάνει ε, με την πηγή, ένα ενεργειακό ε, πόρο για το μέλλον. Το ίτερ που αφορά την ε, σύνδεξη είναι ο γνωστός αντιδραστήρας και όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι 7 ε, οι οργανισμοί που τον χρηματοδοτούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και, και η Ιαπωνία. Αυτή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη τον Απρίλιο. Μία έκθεση δημοσιεύτηκε με βασικά συμπεράσματα, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι επιτέλους ε, δρομολογήθηκε, μπήκε σε μια σειρά αυτό το πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τα πάντα είναι σημαντικά. Ένα νέο πρόγραμμα δράσης, ε, τα οικονομικά ζητήματα, ένα σύνολο θεμάτων λοιπόν ε, και όλη η ενημέρωση που μπορεί να μας δώσει ο Επίτροπος είναι πολύτιμη. Ο κ. Μικελάριας θα πει καλώς ορίζουμε. Η ιδέα συζήτησή μας εντάσσεται στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καμιά φορά σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά για πρώτη φορά συζητούμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις διακοπέ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Με μεγάλη χαρά έρχομαι σήμερα να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για το σχέδιο ITER που είναι από τις μεγαλύτερες συνεργασίες παγκοσμίως σε επιστημονικό τομέα με έξι ευρωπαϊκές χώρες και εκπροσωπούν ε, το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού όπως είπε και η Πρόεδρος. Η βιωσιμότητα και η ασφάλεια φωτιασμού μαζί με την κλιματική αλλαγή είναι βασικά στοιχεία για την ενέργεια ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, αυτές τις προκλήσεις στην Ευρώπη χρειαζόμαστε τολμηρές και καινοτόμες δράσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ήτερ στα λατινικά σημαίνει δρόμος. Είναι πραγματικά μία από τις ε, θαραλέες δράσεις. Ε, Συνένωσε τη διεθνή κοινότητα σε ένα κοινό στόχο και μια κοινή αποστολή να έχουμε καθαρή και απεριόριστη ενέργεια για την καθημερινή μας χρήση. Το σχέδιο ΙΤΕΡ είναι εξέχον, είναι ελπιδοφόρο και ε, μια καταπληκτική λύση που θα μας βοηθήσει να ε, χαράξουμε, να σχεδιάσουμε ξανά τον ενεργειακό χάρτη παγκοσμίω. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σχετικά μεταξύ θέματα κάποιες απόψεις ε, ενεργειακή λύση για αύριο, ευκαιρίες που δίνονται για δημιουργία θέσεων εργασίας και έρευνας ε, για τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή πρόοδος και θα ήθελα να σας αναφέρω και το αναθεωρημένο πρόγραμμα του έργου αυτού. Πάνω από 50% ε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση την εισάγει ως πετρέλαιο κυρίως και φυσικό αέριο από χώρες εκτός της Ένωσης που μπορεί να είναι μακρινές γεωγραφικά ή ασταθείς πολιτικά. Ε, με τις σημερινές τάσεις αναμένεται μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται από ε, εξωτερικούς ε, προμηθευτές για το 70% των αναγκών της. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσει ε, την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία του Παρισίου. Έχουμε νέες δεσμεύσεις για εγκατάλειψη του διοξιδίου του άνθρακα και της οικονομίας του άνθρακα. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα βιώσιμο και ε, με νέες μορφές ενέργειας ανανεώσιμες ε, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε ανεφοδιασμό. Η σύνδεξη ακριβώς αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το καύσιμο είναι απεριόριστο. Ε, δεν επιβαρύνει με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι Εγγενείς, η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν μπορούν ούτε να λιώνουν ούτε να υπάρχουν ε, κάποιες άλλες ε, παράπλευρες απώλειες που υπάρχουν στην σχάση. Ε, και επίσης δεν υπάρχει και θέμα αποβλήτων με μακρά περίοδο ζωής που θα είναι εις βάρος των μελλοντικών γενεών. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το ΊΤΕΡ. Ε, χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις ε, και μέσω αυτής της πύλης θα περάσουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε την εμπορεύσιμη αξία ε, και το κερδοφόρο της υπόθεσης αυτής. Είναι ένα μοναδικό σχέδιο που μπορεί να έρθει σε αίσιο πέρας μόνο με διεθνή συνεργασία χωρών που εκπροσωπούν το μισό πληθυσμό της γης και 80% του ΑΕΠ και οι διεθνείς μας εταίροι ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία χώρα που μπορεί από μόνη της να διεκπαιρέωσει ένα τέτοιο έργο ε, τέτοια ε, διάσταση και τέτοια περιπλοκότητα. Ε, δεν μπορούμε όμω να περιμένουμε δεκαετίε, ούτε χρειάζεται για να δούμε το ωφέλη. Ήδη φαίνονται από σήμερα για τι επενδύσει, την ανάπτυξη και τι εργασίε που είναι και βασικέ προτεραιότητε τη Κομισιόν ενθαρρύνει ε, και τονώνει την ε, ε, επένδυση και την έρευνα των πολιτικών μηχανικών. Δημιουργούνται νέε θέσει εργασία, ιδιαίτερα για μικρομεσαίε επιχειρήσει και νέε επιχειρηματικέ ευκαιρίε, έτσι ώστε γενικά να έρθει η ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην προμήθεια τεχνολογικών στοιχείων και σε 8 χρόνια, από το 2008 ως το 2015, ε, τα ε, ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες έχουν υπογράψει πάνω από 750 συμβάσεις και 150 υποτροφίες έχουν δοθεί ε, αξίας 3,6 δις ευρώ, σχετιζόμενα όλα αυτά με το ΊΤΕΡ. Και πάνω από 300 ευρωπαϊκές εταιρείες και 60 ερευνητικά κέντρα σε τουλάχιστον 20 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ένωσης, συν την Ελβετία, εποφελούνται από την παρούσα επένδυση. Ένα καλό παράδειγμα των ωφελών αυτών είναι η σύμβαση που υπέγραψε τον Ιούνιο η το με μια κοινοπραξία δύο ευρωπαϊκών εταιριών με συμμετοχή και μιας νότιο-κορεατικής. Είναι η μεγαλύτερη σύμβαση ε, του ΙΤΕ, 174 εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση ε, του ΤΟΚΑΜΑΚ, ε, του συστήματος μιας εγκατάσταση που υποστηρίζει. Ένα εκατομμύριο εξαρτήματα πρέπει να συναρμολογηθούν εκεί και καταλαβαίνετε ότι ο Όμιλος και η κοινοπραξία αυτή είναι μια σημαντική επιχείρηση και εγχείρημα. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια πραγματογνωμοσύνη που της επιτρέπει να συνεργάζεται με διεθνείς ε, φορείς και εταιρείε. Επιπλέον, ε, δοκιμάζονται εκεί βασικές τεχνολογίες για το αντιδραστήρα του μέλλοντος στη σύνδεξη. Έχουμε ξεπεράσει ε, την σχάση όπως είναι η μετρολογία, ρομποτική ή η διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι υποστηρίζεται η ε, απασχόληση και η ζήτηση ειδικευμένων εργαζομένων, ε, πολιτικών μηχανικών, ερευνητών και χειριστών προγραμμάτων. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες έμεσες θέσεις εργασίας ε, στη ξενοδοχειακή υποδομή, στον τουρισμό και στην εστίαση στη περιοχή. Μετά την διαδικασία λοιπόν της αρχικής ε, φάσης ε, της συναρμολόγησης θα ακολουθήσει και επόμενη, που και αυτό θα είναι ε, ένα εφαλτήριο για την κατασκευή του εργοστασίου αυτού που θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον του τύπου, όχι μόνο του εξειδικευμένου, αλλά και στον τοπικό και στο διεθνή που παρουσιάζει την πρόοδό του είχε αρχικές δυσκολίες, δεν το κρύβω αυτό, αυξημένο κόστος στην αρχή και καθυστερήσεις από την πρώτη φάση. Αυτό ε, είναι μοιραίο και ε, αναμενόμενο για οποιοδήποτε εγχείρημα τέτοιου μεγέθους. Από το 2015 έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν και να σταθεροποιήσουν ε, οι ενδιαφερόμενοι και τις ε, καθυστερήσεις και το υπερβολικό κόστος. Είναι προφανές ότι προοδεύει ε, εκεί το εργοτάξιο, ιδιαίτερα τα κτίρια που είναι υπό την ευρωπαϊκή ευθύνη. Είμαι βέβαιος ότι Όσοι θα πάτε τον άλλο μήνα στον Κανταράς να επισκεφτείτε το εργοτάξιο θα διαπιστώσετε τη δουλειά που έχει γίνει εκεί. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, έχουν μπει τα θεμέλια ε, για τις οριστικές δράσεις που έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Η οργάνωση ΙΤΕ ενημερώνει τα διάφορα μέρη ε, για την πορεία των εργασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα και νωρίς εντοπίζονται τα ενδεχόμενα προβλήματα και αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις. Τα μισά από τα ορόσημα που έχουν προγραμματιστεί για φέτος έχουν ολοκληρωθεί και ορισμένα αναμένονται προσεχώς. Η διαχείριση της οργάνωσης, η το management, έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να μειώνει τον κίνδυνο. Το τελευταίο Συμβούλιο Ίτερ του Ιουνίου συμφώνησε να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αναθεωρήσεις κρισίμων τομέων του έργου και αποφάσισε ε, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα μέσω ανάλυσης της αποδοτικότητας και ε, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε Και τέλος, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, ε, Έχουμε το Fusion for Energy που είναι η η, μάλλον η σύνδεξη για την ενέργεια ε, που παρακολουθεί και ιδιαίτερα τα θέματα του κόστους και της συγκράτησης αυτού. Τον περασμένο Ιούνιο το Συμβούλιο ΙΤΕΡ ενέκρινε ε, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του σχεδίου ε, μετά την αλλαγή και της διοίκησης το 2015 και στο ΙΤΕΡ και στη δική μας υπηρεσία. Αυτή η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του κόστους είναι πιο ρεαλιστική και θεωρούμε ότι μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ε, είναι η λεγόμενη ε, ημερομηνία για το πρώτο πλάσμα, first πλάσμα και εκεί θα αρχίσει πλέον η λειτουργία. Αυτό τι σημαίνει. Εγκιάτο ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατασκευή του ΙΤΕΡ ε, θα σεβαστεί το ποσό 6,6 δις ευρώ μέχρι το 2020 που είναι η οροφή που έβαλαν οι δημοσιονομικές αρχές το 2010. Με τον χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2020 Βέβαια τώρα αναγνωρίζετε ότι έχουμε ξεφύγει κάπως χρονικά και μπορεί να χρειαστεί επιπλέον πόρους από το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο πέραν του 2020. Παρ' όλα αυτά, το νέο ανεθεωρημένο χρονοδιάγραμμα είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός, διότι μας δίνει ένα σταθερό βήμα, μια σταθερή βάση για πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις με ρεαλιστικό τρόπο. Το νέο χρονοδιάγραμμα βασίζεται σε βαθιά ανάλυση και συστηματικές διαβουλεύσεις με την οργάνωση ITER και τις ε, επιτόπου υπηρεσίες ιδιαίτερα ε, ήταν ε, σημαντική συνεισφορά του δικού μας οργανισμού Fusion for Energy. Μετά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Fusion for Energy αποφάσισε να γίνει ανεξάρτητη αναθεώρηση της δυνατότητας του οργανισμού ε, να ε, συνεισφέρει εγκαίρως ε, στο νέο χρονοδιάγραμμα την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Παράλληλα, συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς στο ITER βάσει της ITER Baseline που αναμένεται να είναι επόμενε φάσει. Από το πρώτο φες πλάσμα στο, στη φάση δευτέριο, τρίτιο κτλ. που αναμένεται και το 2035. Κατόπιν αιτήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων μερών, η οργάνωση ΙΤΕΡ εξετάζει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο να ελαχιστοποιήσει το κόστο χωρί περαιτέρω καθυστερήσει. Αυτό θα παρουσιαστεί το Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει αυτά τα νέα ε, δεδομένα, ιδιαίτερα τα οικονομικά. Σε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο και ε, προετοιμάζει το μέλλον. Μια διάσκεψη σε υπουργικό επίπεδο μάλλον θα λάβει χώρα στις αρχές του επόμενου έτους. Τελειώνω. Το ίτερ είναι ο κρογωνίος των ε, εξελίξεων στην σύνδεξη. Έχουν υπάρξει δραστικές αλλαγές στο έργο, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια που έχουν βάλει τα θεμέλια και γερά θεμέλια για να επιτύχει. Ε, λαμβάνεται υπόψη πλέον η οικονομική δυνατότητα και η έγκαιρη διεκπαιρέωση και ολοκλήρωση των έργων και η λειτουργία του. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη ε, λαμβάνονται υπόψη ανάγκες και απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγαλύτερο μεμονωμένο συνεισφορέα. Οι διεθνεί εταίροι έχουν καταλάβει ε, ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, πέραν των πολιτικών διακηρύσεων θέλουμε να παραμείνουμε ε, η κινητήρια δύναμη αυτού του έργου. Χρειάζονται αλλαγέ, γι' αυτό σα καλώ να συνεχίσετε να υποστηρίζετε αυτή την αναθεωρημένη πρόταση θα πρέπει εγκαίρως να εγκριθεί η νέα βασική γραμμή και να εγγυηθούμε τη χρηματοδότηση μετά από το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο στις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε για αυτήν την ε, ομιλία που είναι πολύ σημαντική και περνάμε τώρα στην ε, συζήτηση με τα μέλη. Ε, συνάδελφοι, θα ήθελα ε, όσοι θα πάρετε το λόγο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων να μην Ορίστε για περισσότερα από 2,5 λεπτά. Αν με επιτρέπετε να σας το ζητήσω. Ο κύριος Ρούμπικ λοιπόν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον ε, Επίτροπο ε, για αυτήν την παρουσίαση. Κατά τη δική μας άποψη το ζητούμενο είναι αυτή η διεθνή συμφωνία και αυτό το διεθνές ερευνητικό έργο που λαμβάνει η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο να ε, εκτελεστεί με επαγγελματικό τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό το εν λόγω ε, σχέδιο προπολογισμού έχει προβλεφθεί για τα επόμενα χρόνια και έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο να τηρηθεί. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν στο επίπεδο της διεθνούς κοινοπραξίας για τις δαπάνε πέρα από το 2020. Δηλαδή, αν τελικά κληθούμε να κάνουμε κάποιε περαιτέρω παραχωρήσει σε επίπεδο δαπανών, ε, πόσο μακριά θα είμαστε διατεθειμένοι να πάμε. Από εκεί και μετά μα είπατε ότι το 50% ε, των οροσύμων ε, μέχρι σήμερα έχουν ε, ε, ολοκληρωθεί, έχουν επιτευχθεί, για μας από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να είχαμε τον λόγο κατάλογο στα χέρια μα, για να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι εκείνα τα έργα τα οποία έχουν επιτευχθεί και ποια είναι τα ορόσημα τα οποία απομένουν για το 2016 και για το 2017, έτσι ώστε το project Fusion for Energy να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε όπως πρέπει νομίζω πως ε, ε, το εν λόγω έργο δεν είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο ε, για την παραγωγή ενέργειας αλλά και ως θεμελιακό project στον τομέα της έρευνας σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό βέβαια θα πρέπει να δώσουμε την κατάλληλη υποστήριξη, να συνεχίσουμε να το υποστήριξουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. νίκα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Κανιέτα, ο οποίος ε, συχνά μας ε, επισκέπτεται για να μας ενημερώσει για τις ε, τελευταίες εξελίξεις. Το γεγονός ότι ε, δίνει τόσο μεγάλη ε, σημασία σε αυτό το project ε, καταδεικνύει ότι πραγματικά τα πράγματα πηγαίνουν όπως πρέπει. Όμως και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες ότι δηλαδή χρειάζεται να συνεχίσουμε τη χρηματοδότησή μας έτσι ώστε να καταδείξουμε το γεγονός ότι συνεχίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση και ότι υπάρχει κάποια προβλεψιμότητα μέχρι σε αυτό το τομέα αλλά όχι απόλυτο. Από εκεί και μετά, εάν θέλουμε να αναλάβουμε ένα ηγετικό ρόλο σε ένα συγκεκριμένο τομέα, ε, τότε ε, ή σε ορισμένου τομεί, τότε ένα από αυτού του τομεί θα πρέπει να είναι ακριβώ αυτό του και θα πρέπει να του δώσουμε την κατάλληλη σημασία. Όχι δηλαδή μέσω των πολιτικών μηνυμάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και μέσω τη χρηματοδότηση των πόρων που δεσμεύουμε. Επίση, ε, να πω ότι θα θέλαμε να, να παρευρεθεί σε κάποια επόμενη ε, συνεδρίαση ε, τη Επιτροπή μα ο Επίτροπο για να μα πει ποιε είναι οι τελευταίε εξελίξει σε σχέση με το πακέτο ενέργεια. σω εκεί λοιπόν σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να μα κάνει μια παρουσίαση για να μα πει ε, ποιε είναι οι κύριε κατευθύνσει στι οποίε κινόμαστε σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ενέργεια, ανανεώσιμε δηλαδή πηγέ ενέργεια, αποδοτικότητα τη παραγωγή ενέργεια και αποδοτικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος για το ECR, το Σενόψικη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Ε, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ε, το ίτερ σε συνδυασμό με τον Καλλιλέο αποτελούν ενδεχομένως τα πλέον σημαντικά ε, τεχνολογικά project τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα δηλαδή μεμονωμένο κράτος μέλος δεν ήταν σε θέση να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο project τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και από άποψη δέσμευση προσωπικού όσο και από άποψη κόστους. Ε, και βέβαια γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση του ΙΤΕΡ δεν ε, μπλέκονται, δεν συμμετέχουν μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το καθιστά ακόμα πιο σημαντικό δηλαδή ακόμα και μετά το 2020 ελπίζουμε ότι θα ε, συνεχιστεί ομαλά το εν λόγω έργο για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε εγκαιρός γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολύ σημαντικές δραστηριότητες ε, σε τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο που απομένουν ακόμα. Δεν έχουν δηλαδή επιληθεί όλα τα ζητήματα σε σχέση με τις συνδέξη και γι' αυτό παρόμοια με τον κύριο Ρούμπι θα ήθελα να ζητήσω και εγώ από τον κύριο Κανέτε να λάβουμε έναν κατάλογο, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο με το τι απομένει, αλλά και με του κινδύνου οι οποίοι ακόμα ελοχεύουν. Γιατί βέβαια κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν σε τέτοιου είδου project. Αν δεν υπήρχαν, τότε δεν θα είχαμε να κάνουμε με ένα τέτοιο πραγματικά πρωταρχική σημασία project. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα πώ θα συμπεριφέρεται το ε, πλάσμα, ποια είναι τα ζητήματα μόνωση σε σχέση με αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν δηλαδή μία σειρά από ε, κίνδυνοι και ερωτήματα ακόμα που παραμένουν να Όπω είπε και ο συνάδελφο, καλό θα ήταν να έχουμε ένα τέτοιο κατάλογο και να έχουμε και τελικά ένα προπολογισμό. Δηλαδή, ποια είναι τα κονδύλια τα οποία τελικά απομένουν, ώστε να στεφτεί με επιτυχία το εν λόγω project. Και να μην δηλαδή ε, αποτύχει με βάση κάποια άλλα ε, διοικητικού χαρακτήρα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ από τη δική μου πλευρά θεωρώ πως είναι πραγματικά εξαιρετικής σημασίας η ενέργεια, η παραγωγή ενέργειας από σύνδεξη, οπότε θα πρέπει να αποτελέσει ένα ε, πρώτη συμβολική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ΙΤΕΝ. Είναι κατά συνέπεια καθήκον μας να ε, παράσχουμε μακροπρόθεσμα ε, χρηματοδότηση αυτό το project. Ναι. η εκ μέρους του Καλημέρα σας κύριε Κανιέτε. Συμφωνούμε απολύτως και εμείς με τη γνώμη σας ότι η σύντηξη ε, θα πρέπει για την Ευρώπη να είναι φάρος, γιατί είναι και μεγάλη οικονομική επιβάρηση αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ μελλοντικά. Η πρώτη ημερομηνία που ακούμε, αν πάνε όλα καλά για εμπορικά αποτελέσματα, θα είναι το 2040. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανανεώσιμες ε, ενέργειες, ε, πηγές είναι οι ε, καθαρές μορφές ενέργειας του παρόντος και όχι του μέλλοντος. Εσείς τι λέτε, για όλα αυτά και αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η μόνη μαζί με την Πορτογαλία και την Ουκρανία, που το 2015 μείωσε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μαραγκάλ, εκ μέρους των Πρασίνων. Α, μόλις μπήκα και θα ήταν άστοχο να τολμούσα να πω το παραμικρό, γιατί δεν άκουσα αυτά που είπε ο Επίτροπος. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς άργησα. Καθυστέρησα και δεν σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. So, Madame, Madame Ernst, as next... Η κυρία Έρνστ, επόμενη ομιλήτρια εξ της Ανατικής Αριστεράς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ακούω αυτά που μας παρουσιάζετε και έχει και μακρά προϊστορία. Το 1951 έγιναν τα πρώτα πειράματα και τώρα είμαστε στο 2016 και δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ έξω και ρωτάω. Τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς. Μιλήσατε για καλό δρόμο, ότι εντάξει πάντα τα πράγματα, έχουμε βελτίωση της διαχείρισης και πολλά άλλα. Τεχνικά από ό,τι διαβάζω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. 100 ε, εκατομμύρια ε, βαθμοί Κελσίου και ότι θα πρέπει κάπως να διατηρείται το πλάσμα σε τόσο υψηλή ε, θερμοκρασία είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα για τη σύνδεξη. Πού βρισκόμαστε, μιλάμε για το 2050 και τέτοιες ε, ημερομηνίες και χρονικούς οριζόντες και το πρώτο πρόβλημα είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Πού βρισκόμαστε, τι είναι ο παραγόν χρόνος εδώ. Και δεύτερον, δεν θα είχε νόημα πολύ περισσότερο να στραφούμε και να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρά σε αυτό το τεράστιο πράγμα που δεν ξέρουμε και τελικά αν μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία. Η κυρία Κάπαλ, εκ μέρου του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Σωστά διαπιστώνετε ότι το ΊΤΕΡ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα του κόσμου τούτου και πολύ σημαντικό φυσικά για τις διεθνείς ε, δικτυώσεις και διασυνδέσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη και η Ευρώπη ως χώρος έρευνας και ανάπτυξης υποφελείται πάρα πολύ, ιδιαίτερα ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με αυτό το Συμβούλιο ΙΤΕΡ τον Ιούνιο κατάλαβε επιτέλους ότι χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα δράσης και ε, χρονικό πρόγραμμα και καλό θα ήταν να το τηρήσει. Ε, σωστό ήταν να αλλάξει και η διοίκηση τον περσινό Μάρτιο έχει καταθέσει το πρόγραμμα δράσης και ε, το Νοέμβριο του 2015 ε, όρισε τους ενδιάμεσους στόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέσσερις από τους έξι αυτούς ε, στόχους ενδιάμεσους του Fusion for Energy έχουν βεβαιωθεί. Καλό σημάδι. Βεβαίως υπήρξαν και στο παρελθόν προβλήματα πολλά και γιατί να το κρύψουμε. Εξού και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αρνήθηκε να δώσει απαλλαγή για το έτος 2014. Στο μεταξύ είχαμε έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουν αυξηθεί κατά 4 δις ε, οι δαπάνες. Έχουμε φτάσει στα 20 δις. Τώρα ακούμε και καθυστέρηση πενταετή για το πρώτο πλάσμα 2025 αντί για 2020. Αλλά γενικότερα έχει σημασία για τη θεμελιώδη έρευνα αυτό. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες σύνδεξης από την DOCAMAC. Υπάρχει το Ινστιτούτο Max Planck που μπορεί σε 19 χρόνια και με κόστος ένα δις ε, να χρησιμοποιήσει άλλη τεχνολογία. Και ήδη παράγεται πλάσμα και πειραματικά. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχουν δυνατότητες ε, να συνεργαστούν το κοιτάνε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΤΕΡ και υπάρχουν και το General Fusion, το 3α Energy στι Ηνωμένε Πολιτείες με κεφάλαια κινδύνου και ιδιωτικά δηλαδή κεφάλαια για να επενδύουν στη θεμελιώδη έρευνα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι κάτι που το σκέφτεστε ε, για το μέλλον, προγραμματίζετε και για το ΙΤΕΡ κάτι τέτοιο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Περνώ το λόγο πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Αριά Κανιέτε, για τη δέσμευση που δείχνει για ένα τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, διότι πρόκειται για ένα διεθνέ ε, πρόγραμμα. Να τον συγχαρώ λοιπόν για αυτή τη μόνιμη του δέσμευση που, με την οποία υπερασπίζεται ένα πρόγραμμα αυτή της εμβέλειας. Δύσκολο όταν ε, γνωρίζουμε πόσο έχουμε αναπόφευκτο αυτή αύξηση των δαπανών, αναπόφευκτη αύξηση όταν προβλέπουμε έργα τόσο μεγάλης διαρκείας, ακόμα και με πολύ προσεκτική διαχείριση, αναγκαστικά ορισμένες δαπάνες δεν ε, μπορούν να προβλεφθούν ε, με απόλυτη ακρίβεια. Ευχαριστούμε λοιπόν. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα διεθνέ πρόγραμμα θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι ο μεγαλύτερο χρηματοδότη, 45% αν δεν απατώμε, 45,5% αλλά μάλιστα ο αντιδραστήρα θα βρίσκεται επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Πέραν αυτού του προγράμματος σύνδεξης, όλα αυτά απαιτούν νέες επιστημονικές τεχνολογικές γνώσεις και που θα εξυπηρετήσουν και πολλούς άλλους βιομηχανικούς τομείς. Έχουμε πολλοί αριθμούς εταίρους ανά τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Ινδία. Ήθελα να μου πείτε, πώς βλέπετε τις θέσεις των διεθνών μας εταίρων. Είναι εξίσου ενθουσιασμένοι, έχουν την ίδια ισχυρή βούληση όπως εσείς κύριε Επίτροπε να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα και φυσικά να δεχθούν και ε, τις τυχαίες ε, περιπλοκές που μπορεί να συνεπάγεται ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επίτροπη συχνά είναι ευέλικτη, αλλά η βουλευτέ είναι ευελικτοί και επειδή έχουμε κάποιε πολύ σημαντικέ ε, εκκρεμότητε ενώπιον μα για τι επόμενε δύο εβδομάδε, θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να θέσω ένα σχετικό ερώτημα. Μέσα στι επόμενε ε, ημέρε, ε, κύριε Επίτροπε, θα υποβάλλετε την αναθεώρηση για τη νέα οδηγία, για την αναθεώρηση τη οδηγία την εφαρμοστική λοιπόν έκθεση και με βάση κάποια στοιχεία που είχε υπολογίσει η Επιτροπή ως το 2020, Ε, δεν θα επιτύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει για, έως το 2020 για λίγο σε ό,τι αφορά την ε, αποδοτικότητα. Υπάρχει όμως ε, ε, ένα άλλο ε, υπόμνημα της Επιτροπής ε, η οποία αναφέρεται στο ότι ήδη από το 2014 έχουμε επιτύχει αυτήν την, τον, το στόχο της ενεργής αποδοτικότητας. Αυτό είναι εντελώς παράδοξο. Δηλαδή η έκθεση που είχαμε λάβει είναι εντελώς εσφαλμένη και ποιες είναι τελικά οι συνέπειες από αυτό. Θα αναβάλλεται την ε, εξέταση, την αξιολόγηση της ε, εφαρμογής ε, της οδηγίας για την ενεργή βιωσιμότητα ή όχι. Τι ακριβώς θα κάνετε σε σχέση με αυτό. Στο πολύ κύριε συνέδριο, κύριος Μπενίτος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, όταν μας μιλάτε για το σχέδιο ΙΤΕΡ, είναι σαν να μας μιλάτε για κάποιο μαγικό ραβδάκι που θα εξασφαλίσει τον εφοδιασμό, θα σταματήσει την κλιματική αλλαγή, θα λύσει την ενεργειακή φτώχεια και την ανεργία. Κάπως έτσι μας είχαν παρουσιάσει στην αρχή την ηλεκτρική ενέργεια. Και στις δύο περιπτώσεις αναπαράγεται το μύθος ότι έχουμε ανεφοδιασμό ανεξάντλητο. Ε, ωστόσο, και ας υποθέσουμε ότι θα ε, ε, λύσουμε τους αγνώστους χείρι της τεχνολογίας του έργου. Μήπως έχουμε πάρει το δρόμο παραγωγής ενέργειας πολύ πιο επικεντρωμένης και συγκεντρωτικής και οικονομικά και γεωγραφικά ακόμα περισσότερο γίνεται αυτό και μακριά από την κατανάλωση, άρα πιο ανεποτελεσματική. Και πού είναι ο, ο καθαρός χαρακτήρας, είναι σχετικός κατά την άποψή μας. Όπως και τα συμβατικά πυρηνικά εργοστάσια, μόλις τελειώσει ο χρόνος του, ο λειτουργικός, θα πρέπει να διαλυθεί, να παροπλιστεί αυτό, που θα είναι μετά από 39 χρόνια και μάλλον παράκριβο, περίπου 40 χιλιάδες τόνους ε, ραδιενεργά μέταλλα θα έχουμε να πετάμε από τότε. Και τι θα το κάνουμε αυτά. Σε άγνωστο μέρος θα αποθηκευτούν. Έχω λοιπόν μια αφιβολία, κύριε Επίτροπε. Τα γνωρίζετε όλα αυτά ή τα σκέφτονται, τα, τα μελετάτε. Ποιος θα, ε, είναι ε, ο τελικός στόχο, τελική τιμή της κιλοβατόρας και ε, αν σήμερα θα συνυπολογίζετε και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Εδώ ολοκληρώθηκε ο κατάλογος ομιλητών. Θα θέλαμε τώρα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το πρόγραμμα αυτό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο περισσότερες ερωτήσει μπορώ. Να πω στον κύριο Ρούμπικ και στους λοιπού ομιλητέ πρώτα απ' όλα. Μέχρι στιγμής κυρία Γκροστέτα, η δέσμευση όλων των μερών ε, του ΙΤΕΡ ε, υπογραμμίστηκε ξανά στο Συμβούλιο του Απριλίου του 2016. Κάθε μέρος, χώρα μέρος του ΙΤΕΡ, επικύρωσε τη συμμετοχή του στον προπολογισμό του οργανισμού ΙΤΕΡ. Εφόσον λοιπόν διατηρείται το ενδιαφέρον των μερών για τη σύνδεξη, ενδιαφέρονται και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, διότι σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να κατασκευάσει και να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα τέτοιας εμβέλειας και τέτοιου είδους. Θα θυμάστε ε, ότι παλιότερα όταν εμφανίστηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν ήταν σαφείς οι αρμοδιότητες. Ε, τώρα λοιπόν είναι σαφώς υπό τη δική μου αρμοδιότητα και το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι ε, να έχουμε καθαρή ε, διαχείριση του προγράμματος, τη διοίκηση και τώρα έχουμε τον οργανισμό. Έχουν γίνει και οι αλλαγές στον οργανισμό ΙΤΕΡ που εισήγαγε η νέα διοίκηση βάσει του διαχειριστικού σχεδίου της και κυρίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού ΙΤΕΡ και των ε, οργανισμών της κάθε χώρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι βελτιώθηκε ο τρόπος εργασίας μας. Δεύτερον, ε, δημιουργήσαμε ένα χρονοδιάγραμμα από κοινού στον οργανισμό ΙΤΕΡ και από τους εγχώριου οργανισμούς. Για πρώτη φορά έγινε κάτι τέτοιο από κοινού, ενώ φαίνεται κάτι λογικό. Πρώτη φορά συνεργάστηκα μεταξύ τους για να καθορίσουν την προσέγγιση η οποία επικυρώθηκε και από ανεξάρτητους ε, ελεκτές και η υλοποίηση αυτής της προσέγγισης θα υποστηριχθεί από αυτή τη διοίκηση βάσει κάποιων, ε, μιας, ενός ολοκληρωμένου καταλόγου οροσίμων, βάσει των οποίων μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο. Τα ορόσημα ε, που ορίστηκαν τον Νοέμβριο του 2015 από το Συμβούλιο έχουν προχωρήσει πολύ. Πάνω από το 15% έχει επιτευχθεί, όπως είπα. Θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες, αφού μου ζητήθηκε να δώσουμε τον κατάλογο των ε, έργων. Θα σας δείξουμε τι έχουμε επιτύχει, ποια έργα έχουν υπάρχουν στο τραπέζι. Με ρώτησαν για τις ημερομηνίες. 2025 για το πρώτο πλάσμα, 2035 για την δραστηριοποίηση. Το συνολικό ποσό ε, συμμετοχών σε χρήμα και σε είδος. Σε χρήμα η συμμετοχή που απαιτείται για την κατασκευή από όλα τα μέρη για την περίοδο 2016-2025 εκτιμάται από τον ορισμό ΙΤΕΡ σε περίπου 5,5 δις ευρώ ε, αξίας 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, όπως υποθήκατε πολύ σωστά, θα πληρώσει το 45% αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί επίσης να ε, συμβάλλει και σε είδο σύμφωνα με τη συμφωνία ΙΤΕΡ. Η συμμετοχή λοιπόν ε, σε είδο επηρεάστηκε από το νέο χρονοδιάγραμμα. Οπότε πρέπει να επανυπολογιστούν. Και αυτή τη στιγμή η Φυσιοφρονέζη ε, προετοιμάζει τις εκτιμήσεις των συμμετοχών αλλά σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν εντός των ορίων που έχουν οριστεί για το πλαίσιο και μόλις έχουμε τα δεδομένα θα σας τα δώσουμε για το 2025 και η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μια πολύ λεπτομερή ανάλυση για να λάβει την εγκρίση της Δημοσιονομικής Αρχής με το νέο κόστος κατασκευής και επίσης για την έγκριση της νέας βάσης του προγράμματος. Σύντομα θα τα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Νομίζω τον Νοέμβριο. Μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση. Τον Νοέμβριο φέτος θα είμαστε σε θέση να σας τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Ε, κυρία Πονσέτ, πότε θα δεθεί σε λειτουργία το 2035. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα 2040. Ρωτήσατε τι γίνεται με τις ανανεώσιμες στην Ισπανία. Και στην Ισπανία και παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας είναι ο στόχος, 20% για τις ανανεώσιμες. Και έχουμε και ένα μονοπάτι που έχουμε πάρει και ε, ένα σύνολο ανανεώσιμων, το πρόβλημα και το μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να φτάσουν 27 σε μία χώρες στο στόχο αυτό. Το, την Άνοιξη θα δημοσιεύσουμε τα νέα κλειστά στοιχεία να δούμε πού βρίσκονται τα διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ανανεώσιμες πήγες δεν είναι μόνο ε, η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή, είναι και η βιομάζα. Και στην Ισπανία και σε πολλά κράτη-μέλη. Αν ε, τα προσθέσουμε ε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ε, η βιομάζα δεν συνομπολιγιζόταν γιατί δεν υπήρχαν τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας. Τώρα που ξέρουμε τι στοιχεία μπορούμε να προσθέσουμε, να αθροίσουμε, θα δούμε τι συμβαίνει στα κρατημέλη και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε όλοι να φτάσουν στο στόχο. Ακούσαμε για την ενεργειακή απόδοση και για το ότι θα σας προτείνουμε ως δέσμες και μέτρα. Κοιτάξτε, το πιο περίπλοκο ίσως από πλευράς εκτέλεσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η ενεργειακή απόδοση. Energy efficiency στα αγγλικά. Ε, αυτά είναι από τα πιο δύσκολα και εκεί τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερες δυσκολίες σε πολλούς τομείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκινεί διαδικασίες επί παραβάση για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό στην ε, εθνική τους νομοθεσία, δεν τα έχουν μεταφέρει δηλαδή. Τι άλλο ε, με ρωτήσατε. Uh, Μια περίπλοκη ερώτηση έκανε ο κύριος Σουλουάγκα για το πώς υπολογίζουμε το κόστος ε, παροπλισμού. Μα τώρα εμείς το χτίζουμε από την αρχή αυτό το εργοστάσιο, αυτή την εγκατάσταση. Μετά δεν θα είναι υπερβολικά συγκεντρωμένο. Τώρα έχουμε ε, ένα ενιαίο χώρο, αλλά για το είναι. Ε, εμπορική δραστηριότητα θα έχουμε άλλες μονάδες πιο μικρές, αποκεντρωμένες. Και επίσης έχουμε κάποια εμπειρία με παροπλισμό πυρηνικών ε, εργοστασίων. Μπορούμε να υπολογίσουμε με σχετική ακρίβεια ε, Τρία είναι τα project που υποστηρίζουμε ήδη με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ξέρουμε Εξάντε εκ των προτέρων δηλαδή ποιο θα είναι το κόστος. Τώρα μιλάμε για διαφορετικό καύσιμο επίσης και θα είναι διαφορετική και η διάθεση των αποβλήτων. Πάντω έχει βάσει αυτή η ιδέα ότι να μην σκεφτόμαστε μόνο την τεχνολογία αλλά και πώ θα γίνει ο παραπλησμός, η διάθεση των αποβλήτων και βεβαίω αυτά τα σκεφτόμαστε και μα απασχολούν. Επίση, ακούσαμε κάποιε ερωτήσει ε, γιατί ε, υπάρχει υποστήριξη από πολλά κράτη. Είναι ένα μοναδικό έργο. Αν δεν υπήρχε η υποστήριξη των κρατών και από τους δημόσιους ε, προϋπολογισμούς θα ήταν αδύνατον να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, το να δημιουργηθούν αυτή η υποδομή, το να υπάρχει η συμβολή σε χρήμα και σε είδος, ε, να υπάρξει η συνεργασία με τον τομέα. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχαμε επίσης συστήματα υποστήριξης, ε, δασμολογικές ευκολίες, ε, διάφορα στοιχεία τα οποία προσέλξαν τον ιδιωτικό τομέα και τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνονται ανταγωνιστικέ αυτέ οι ανανεώσιμε μορφέ ενέργειας χωρίς δημόσια στήριξη. Ενώ αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα χρειαστεί τη δημόσια στήριξη για να αναπτυχθεί. Και το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια σαφή εικόνα του κόστου. Έχουμε μια ε, πολιτική δημοσιονομική προοπτική μέχρι το 2020 θα είμαστε εντό των ορίων. Είναι σαφέ ότι μετά από το 2020 στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική θα χρειαστεί αύξηση από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, των συστημάτων υποστήριξης προ τα ε, κράτη-μέλη. Μετά ρωτήθηκε αν υπάρχουν και παράλληλες καινοτόμες τεχνολογίες. Εμείς αναπτύσσουμε αυτήν. Έχουμε τα πρόγραμμα Horizon 2020 και μετά θα έχουμε το διευρυμένο σχέδιο Juncker, όπου υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία που σχετίζεται με την κλιματική δράση και τις, ε, ενέργειες, τις μορφές ενέργειας του μέλλοντος, οπότε εκεί θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και άλλων ε, προγραμμάτων. Το παράθυρο αυτό, το περιθώριο αυτό είναι 40% των διαθέσιμων κονδυλίων για κλιματική δράση, καθαρή ενέργεια και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδος ενέργειας που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα υποστηρίξει την επιτεύξη των στόχων μας. Έχουμε χρηματοδότηση για αυτά. Τώρα, αυτό που θέλω να πω σε αυτήν εδώ την Επιτροπή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα αυτό και συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Συμμετείχαμε στην εκλογή του νέου ε, Γενικού Διευθυντή, ε, στην κατάρτιση των σχεδίων δράση. Το παρακολουθούμε καθημερινά και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Που πάει κανεί εκεί, βλέπει πώ λειτουργεί, κάνει όλε τι ερωτήσει και πηγαίνετε εκεί εσείς και μετά μας λέτε τι εντύπωση σας έκανε. Ε, μας αρέσει που θα πάτε εκεί, δηλαδή να λάβετε πληροφορίε, αλλά θέλουμε να δούμε και τι βλέπετε κι εσείς. Είναι εντυπωσιακό. Είναι κάτι μοναδικό. Και είναι εντυπωσιακή η ποιότητα. Τώρα έχουμε τα δοχεία πίεση τα δοχεία κενού και οι Κινέζοι δουλεύουν τους μαγνήτες. Ε, είναι ε, κάτι μοναδικό. Και λέμε ότι είναι ναι, μια λύση καθαρή ενέργεια. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια ε, μίζωνο σημασία καινοτομία, διότι θα μπορούμε να παράγουμε καθαρή ενέργεια με πολύ χαμηλότερο κόστο και να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ούτε την ενεργειακή απόδοση, ούτε του κλιματικού μα στόχου. Κάνουμε τα πάντα ταυτόχρονα. Η Κομισιόν ε, έχει δεσμευτεί πραγματικά και αφοσιωθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξουμε το ταχύτερο δυνατόν το ενεργειακό μας μείγμα, παράγοντας ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναπτύσσοντας ε, συσσωρευτές, ε, χώρους αποθήκευσης, ε, φέτος ε, θα εμφανιστούν και η σχετική νομοθεσία ώστε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους ενεργειακούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν θα έχουμε λοιπόν τις σχετικές οδηγίες ε, και τη σχετική νομοθεσία, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να εμφανιστεί πρώτη και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων είναι το μόνο που θα περιμένει λίγο. Το Μάρτιο ήδη λοιπόν του χρόνου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει όλη την απαραίτητη νομοθεσία για την επιτεύξη των κλιματικών μας στόχων. Προς εξέταση. Ευχαριστώ, πολύ. Κύριε Επίτροπε. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Τα η ημερομηνία που θα τελειώσει τώρα αυτό έργο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, απαντηθεί αυτό το επιστημονικό έργο, επίσης τα χρήματα που θα χρειαστούν στην Επιτροπή μας είμαστε πεπισμένοι για ε, το εγχείρημα αυτό, οι περισσότεροι από εμά. Δεν χρειάζεται να μας πείσετε. Ίσως να μην συμβαίνει το ίδιο στο υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και κάτι άλλες. Αλλά εδώ στη δική μας Επιτροπή δεν χρειάζεται, έχετε πολλούς υποστηρικτές και ένθερμους. Ιδιαίτερα στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, σας το λέω και θα σας σταλεί ιδιαίτερη ενημέρωση, έχουμε ειδική ε, αποστολή εκεί για να τα δούμε ειδή σώμαση. Αν ενδιαφέρονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, μπορούμε να διοργανώσουμε και μια δεύτερη επίσκεψη λίγο αργότερα. 24 Οκτωβρίου, λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, του Στρασβούργου, να Είστε έτοιμοι. Ε, Στι 23 του μηνό θα πρέπει να είστε την Κυριακή εκεί, στο Καταράς. Ε, δεν ξέρω, ίσως να έχουμε συζητήσεις ε, το βράδυ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μπορούμε να ρωτήσουμε και τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πολλοί έχουν ξεσηκωθεί και λένε ότι δεν χρειάζεται άλλα λεφτά για το ίτερ. Η Επιτροπή ίτερ όμως, η δική μας, είναι στο πλευρό σας και παρακαλώ τους συναδέλφους μην διστάσετε να δηλώσετε 24 ε, Οκτωβρίου στις 23 να είμαστε επιτόπου και τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαστε στο Στρασβούργο. Μπορείτε και να υπογράψετε δηλαδή στο Στρασβούργο. Τα έχουμε σκεφτεί όλα και τα έχουμε όλα προετοιμάσει και φροντίσει. Μπορείτε και το είτε να επισκεφτείτε και το βράδυ να είσαστε στο Στρασβούργο με απευθείας πτήση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Και σας ενθαρρύνω όλους να δείξετε ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνάδελφοι, στις 12 και 13 Οκτωβρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, πρωί και απόγευμα. Είναι τέσσερις μήνες σύνοδοι, δύο μέρες, τέσσερις μισές μέρες. Και στις 14 συνεδριάζουν οι συντονιστές. Πολλές συζητήσεις. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Επίτροπε. Γεια σας.